Καλησπέρα σε όλους. Καλωσορίζω τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων που συμμετέχουν στη Διακοινοβουλευτική Επιτροπή. Η σημερινή συνεδρίαση διαιρείται στα δύο. Πρώτο μέρος. Ψηφιοποίηση και το μέλλον της, το μέλλον της εργασίας. Δεύτερο μέρος, ανισότητες στα κράτη-μέλη. Πριν μπούμε στην ουσία των συζητήσεων, να κάνω κάποιες ανακοινώσεις. Έχουμε κάρτες για εκείνους που θέλουν να πάρουν το λόγο, να συμπληρώσετε τις κάρτες αυτές και να τις δώσετε αν θέλετε να λάβετε το λόγο. Οι λευκές κάρτες αγορεύσεων είναι για το πρώτο τμήμα της συνεδρίσεως και οι κίτρινες για το δεύτερο θα έχουμε την εξή υποδιέρεση τη χρονική. Θα ακουστούν τρει εθνικοί βουλευτέ στη σειρά, μετά θα ακολουθήσει ένα ευρωβουλευτή, θα πάρει το λόγο, μετά άλλοι τρει εθνικοί βουλευτέ και το καθεξη καθεξή. Τρία-ένα, τρία-ένα. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, ε, είμαστε έτοιμοι είμαστε και ευέλικτοι από αυτόν. Να πω κάποια πράγματα εν είδη εισαγωγή για το πρώτο μα θέμα δηλαδή η ψηφιοποίηση και το μέλλον της εργασίας. Κυρίες και κύριοι, το μέλλον της εργασίας ή το, η εργασία του μέλλοντος. Μας χτυπάει την πόρτα. Δεν απέχει και πολύ, παρόλο που υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες ε, ασαφείς. Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Η ψηφιακή οικονομία, η ψηφιακή αλλαγή θα μεταμορφώσει την αγορά εργασίας. Και δεν θα υπάρχει πλέον περιθώριο για επαναλαπτικές εργασίες χαμηλών δεξιοτήτων θα αντικατασταθούν μερικώς από αυτόνομα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Και γι' αυτό υπάρχουν πολλές ανησυχίες και πολλοί φόβοι που περιστρέφονται γύρω από την αλλαγή. Σύμφωνα με διάφορες έρευνες, τουλάχιστον 65% των σημερινών θέσεων εργασίας στην Ευρώπη θα επηρεαστούν από αυτές τις εξελίξεις. Οι γραμματιακές θέσεις, ε, ανειδίκευτοι εργάτες, μηχανικοί οδηγοί, εκείνοι που χειρίζονται μηχανήματα θα αντικατασταθούν κατά 60-80%. 10 με 15% των θέσεων εργασίας των σημερινών θα εξαλειφθούν σε μερικές ε, δεκαετίες. Και αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική καμπή σε σχέση με τις παλιές βιομηχανικές αλλαγές, όπου 4 με 5% των θέσεων εργασίας θα είχαν απολεστεί και θα είχαν αντικατασταθεί. Υπάρχουν όμως και καλές ειδήσει. Και χάρη στον αυτοματισμό και στη ρομποτική αρχίζουν και εμφανίζονται νέες μορφές εργασίας, ενδιαφέρουσες, όσον αφορά τη δημιουργικότητα και τη διάδραση με τα μηχανήματα. Αυτές είναι οι αυριανές ε, θέσεις εργασίας και γι' αυτό αναφερόμαστε στην τέταρτη βιομηχανική ε, επανάσταση που είναι η ψηφιοποίηση της οικονομίας. Βέβαια τα κράτη-μέλη είναι σε διαφορετικά επίπεδα όσον αφορά αυτή την επανάσταση. Στη χώρα μου μόλις τώρα αρχίζει, αλλά η καλή παιδεία θα είναι το κλειδί της επιτυχίας αυτήν την οικονομία. Πάνω από 10% των εργοδοτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια θα χρειάζονται καλά εκπαιδευμένο προσωπικό με πολλά προσόντα και βέβαια ψηφιακή τεχνολογία, η ε, τεχνογνωσία, οι διάφορες δεξιότητες στο διαδίκτυο θα έχουν μεγάλη ζήτηση. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ε, οι δουλειές οι ανθρώπινες θα χαθούν. Όλα θα είναι θέμα διάδρασης μεταξύ ε, των παλιών θέσεων και των νέων θέσεων. Σε ένα πνεύμα πραγματισμού ελπίζω ότι σήμερα θα τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα και θα προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιες απαντήσεις ε, πριν καν σκεφτούμε τη θέσπιση κανονισμών για τη μελλοντική νομοθεσία, ίσως μπορούμε να σκεφτούμε κάποια μελλοντικά επιχειρηματικά μοντέλα, τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, συλλογικές διαπραγματεύσεις, κοινωνικό διάλογο κλπ. Και θα υπάρξει ένα νέο είδος ψηφιακού εργαζομένου που θα έχει διάφορες διεξόδους για να μπορεί να ε, ολοκληρωθεί επαγγελματικά ανάλογα με την ε, τεχνολογία που θα είναι διαθέσιμη. Θα πρέπει να διαρωτηθούμε ποιο θα, ποια θα είναι η μορφή αυτού του μελλοντικού ψηφιακού εργαζόμενου που η δουλειά του μόνο υποβοηθείται από ψηφιακά μηχανήματα ή από κάποιο εργαζόμενο που είναι ειδικό για την πληροφορική και μπορεί να διαμορφώσει το ρομπότ ή το μηχάνημα το ψηφιακό, να το προγραμματίσει. Τι γίνεται για το εργατικό δίκαιο έχουμε τον, εργοδότη και τον εργαζόμενο σήμερα. Θα ισχύει και αυτό αύριο. Θα πρέπει να εισαγάγουμε νέες νομικές έννοιες που θα λαμβάνουν υπόψη το νέο περιβάλλον εργασίας. Και θα πρέπει οι εργαζόμενοι να έχουν ένα επαρκές επίπεδο προστασίας. Θα πρέπει να σκεφτούμε ποιες είναι οι συνέπειες της ψυχιακής οικονομίας, συνέπειες για την ίδια την νομοθεσία και σε ποιο βαθμό θα μπορούμε να νομοθετούμε το περιβάλλον το εργασιακό το αυριανό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εθνικές κυβερνήσεις και οι κοινωνικοί εταίροι ήδη ξεκίνησαν συζητήσεις ούτως ώστε να καθορίσουν το πολιτικό θεματολόγιο και το νομικό θεματολόγιο για το κατάλληλο επίπεδο προστασίας ε, για τους εργαζόμενους. Αυτή η διάσκεψη είναι ένα κομμάτι της όλης προσπάθειας. Η χώρα μου προεδρεύει του Συμβουλίου για το εξάμεινο αυτό και διοργάνωσε αυτή τη διάσκεψη για το μέλλον της εργασίας βάσει της ε, όλης ε, προσέγγισης του κύκλου ε, ζωής. Θα γίνει στη Σόφια η διάσκεψη και θα συζητηθούν εκεί όλα αυτά τα θέματα, η απασχόληση σε σχέση με την ψηφιοποίηση και ελπίζουμε ότι θα ε, καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα στη διάσκεψη και ότι αυτά τα συμπεράσματα θα ληφθούν υπόψη σε συμπεράσματα του Συμβουλίου προς υιοθέτηση τον Ιούνιο. Σας συμπρόεδρος της σημερινή διασκέψεως, ελπίζω ότι θα είναι χρήσιμη η συζήτησή μας και το όλο εγχείρημα θα είναι ενδιαφέρον και χρήσιμο. Αν θέλετε, δίνω το λόγο στην κυρία Μαρίτα Ουλσκογκ, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας, Απασχόλησης και Κοινωνικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Χαρά για μένα να παρίσταμε και που παρίσταστε. Σας καλωσορίζω για τη διακοινοβουλευτική αυτή συνεδρίαση. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο αυτό το ζήτημα, όπως και σε άλλες χρονιές. Λαμβάνεται υπόψη στην Ευρωπαϊκή, λαμβάνει χώρα στην ε, διακοινοβουλευτική Ευρωπαϊκή Εβδομάδα. Συμμετέχουν ε, βουλευτές από την Ευρωπαϊκή Ένωση να συζητήσουν θέματα που είναι πολύ σημαντικά για όλους μας και για το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Χαίρομαι που σημειώνω που πάνω από 245 βουλευτές συνολικά θα παραστούν αυτή την εβδομάδα σε διάφορα σεμινάρια, σε διάφορες ακροάσεις. Έχουμε πολλές τέτοιες εκδηλώσεις και πάνω από 33 βουλευτές συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση από 22 κράτη-μέλη. Θα συμμετάσχουν λοιπόν σε διάφορα τμήματα των συζητήσεων ή σε ολόκληρη την συνεδρίαση. Έχουμε λοιπόν μια άκρο ενδιαφέρουσα εισαγωγή που έγινε στο θέμα της ψηφιοποίησης. Πολύ σημαντικό θέμα, 65% όπως είπε και ο Σαντίμοφ, 65% της αγοράς εργασίας θα αλλάξει, θα μεταλλαχθεί μέσω ψηφιοποίησης και ίσως και μεγαλύτερο ποσοστό. Και όχι μόνο η αγορά εργασίας θα αλλάξει, αλλά η κοινωνία, η δημοκρατία, η καθημερινή μας ε, ζωή θα επηρεαστεί. Τεράστιο θέμα που πρέπει να συζητήσουμε θα δώσουμε το λόγο τώρα στον επόμενο ομιλητή. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν την κυρία Ούλσκοκ για τα εισαγωγικά της σχόλια και θα ήθελα να μου επιτρέψετε αγαπητοί συνάδελφοι να δώσω το λόγο στον κύριο Χένρικ Μπόγκαρτ που είναι από την Βελγική Βουλή το λόγο για 8 λεπτά για να μας κάνει και αυτός με τη σειρά του μια παρουσίαση. Inclusive economic growth emphasizes Θα ήθελα λοιπόν να μιλήσω για την ψηφιοποίηση των οικονομιών μας και για τον τρόπο με τον οποίο μεταλλάσσεται ο κόσμος της εργασίας. Στην εισαγωγή που θα κάνω σε αυτό το περίπλοκο θέμα θα ασχοληθώ με κυρίως δύο σημεία. Πρώτα απ' όλα τη δημιουργία ε, και την απώλεια θέσεων εργασίας που δημιουργεί η ψηφοποίηση και δεύτερον την εκπαίδευση και τις δυνατότητες που δίνονται μέσω της παιδείας. Να σας πω πως η αλλαγή μέσω ψηφιοποίησης ενέπνευσε και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός για να καταλήξει στα εξή συμπεράσματα. Καταρχήν, η ψηφιοποίηση θα μπορούσε να δημιουργήσει μέχρι το 2025 6 εκατομμύρια θέσεις εργασίας παγκοσμίω στα logistics και στα ηλεκτρονικά. Σε άλλους κλάδους όμως η αυτοματοποίηση θα μειώσει κατά 200 εκατομμύρια μέχρι 2 δισεκατομμύρια θέσεις εργασίας μέχρι το 2030. Βλέπετε λοιπόν πως είναι πολύ μεγάλο το φάσμα και η συζήτηση σε πολιτικό επίπεδο δεν ε, ξέρουμε πού θα οδηγηθεί. Επίσης υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα για τους μισθούς, για τις συνθήκες εργασίας προκύπτει το εξή θέμα. Πώς μπορούμε με ενεργητικό τρόπο να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που θα εμφανιστούν. Θέλουμε στεναρή ηγεσία που θα χαράξει το δρόμο έτσι ώστε να έχουμε ένα βιώσιμο πλαίσιο για τα μεμονωμένα άτομα και για τις επιχειρήσεις μέσα σε αυτό το καινούργιο μοντέλο. Έτσι ώστε να αγκαλιάσουμε τη νέα ψηφιοποιημένη ε, οικονομία για τους επόμενες γενναίες και αυτό πρέπει να το κάνουμε ήδη σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2018. Είμαστε μια ένωση αξιών και εδώ πρέπει να λάβουμε τις θεμελιώδεις αποφάσεις έτσι ώστε να μην αφήσουμε κανέναν πίσω. Είτε είναι επιχείρηση, είτε είναι με μονομένους εργαζόμενους. Μία λοιπόν στρατηγική που θα συμπεριλαμβάνει όλους με νέες ε, ευκαιρίες και με νέα μοντέλα, έτσι ώστε να αποφύγουμε τον αποπληθωρισμό, τις κοινωνικές αναταραχές και να προετοιμαστούμε καταλήλως για το ψηφιακό μέλλον. Σύμφωνα με τις έρευνες που έχει κάνει το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, έχουμε τρεις κατηγορίες ε, θέσεων εργασίας που χωρίζονται σύμφωνα με πολλούς ε, συγκεκριμένους παράγοντες. Καταρχήν, η μάχη κατά των μηχανών. Έχουμε εδώ το διοικητικό προσωπικό, έχουμε τους οδηγούς φορτηγών, ε, έχουμε θέσεις οι οποίες θα εξαφανιστούν. Έχουμε αυτούς που τρέχουν με τη μηχανή, δηλαδή για τους ε, χειρουργούς για παράδειγμα, που χρειάζονται κάποιες δέτερες δεξιότητες και μια τελευταία κατηγορία, αυτοί που τρέχουν γρηγορότερα από τη μηχανή ή τρέχουν σε άλλο αγώνα. Είναι οι νέες θέσεις εργασίες, οι δημιουργικές ε, τέχνες, η διαχείριση δεδομένων και μηχανών. Λοιπόν, Παρ' όλα αυτά, η επιπτώση τη ψηφιοποίηση ξεπερνά τα απλά εργασιακά θέματα, γιατί θα αλλάξουν τελείως οι κοινωνίες μας μέσα στις επόμενες δεκαετίες. Αγαπητοί συνάδελφοι, εμείς εδώ μιλάμε για τις ευκαιρίες που μπορούν να προσφέρουν αυτές οι νέες τεχνολογικές δυνατότητες. Βέβαια αυτά δεν θα συμβούν αυτόματα ούτε με τόσο διαστρωμένο τρόπο ούτε πάντα προ όφελο τη κοινωνίας. Θα πρέπει όσοι λαμβάνουν πολιτικές αποφάσεις να αντιμετωπίσουν κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα για τα εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να στρέψουμε την βιομηχανία προς τέτοιου είδους ψηφιοποιημένα εργαλεία προς όφελος της κοινωνίας, μειώνοντας τα εμπόδια για τις επιχειρήσεις με πραγματική παγκοσμιοποίηση όλων των κλάδων. Η ψηφιοποίηση μπορεί να φέρει κοινωνικο-οικονομικά πλεονεκτήματα. Είμαι πεπισμένο γι' αυτό και στην ανάλυση των επιπτώσεων, στην ανάπτυξη και στην απασχόληση, η Price Waterhouse καταλήγει το να δημιουργήσουμε ψηφιακές αγορές μπορεί να αποδώσει ιδιαίτερα οικονομικά ωφέλη και να οδηγήσει σε σημαντικά κοινωνικά ωφέλη για τις κοινότητες και τις κοινωνίες. Και δεν θα πρέπει να υποεκτιμήσουμε τον κίνδυνο της ε, απώλειας θέσεων εργασίας. Για ένα μεγάλο κομμάτι της απάντησης μπορεί να φαίνεται απλοϊκό, παιδεία κατάρτιση, αλλά χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια από όλους, γιατί ολόκληρες ομάδες της κοινωνίας μας θα πρέπει να κινητοποιηθούν εάν θέλουμε να επανεκπαιδευτούν έτσι ώστε να ωφεληθεί και ο επιχειρηματικός κόσμος αλλά και η κοινωνία έτσι ώστε να ανοίξουν ορίζοντες στους οποίους δεν γνωρίζαμε στο παρελθόν. Η πολιτική συζήτηση θα πρέπει να ξεκινήσει από το πώς μπορούμε να μοιράσουμε τα πλεονεκτήματα της αύξησης της παραγωγικότητας. Σε μια κοινωνία ανοιχτή σε όλους θα πρέπει, είναι προφανές, να επενδύσουμε στην παιδεία έτσι ώστε κάθε μέλος της κοινωνίας να εκπαιδεύεται, να επιμορφώνεται, να καταρτίζεται για να παραμένει ενεργό μέλος αυτής Διαφορετικά πώς μπορούμε να ζητήσουμε από ανθρώπους να σέβονται τους κανόνες και τις παραδόσεις αν η κοινωνία δεν τους σταθεί τη στιγμή που την χρειάζονται περισσότερο. Θα πρέπει επίσης να ξεπεράσουμε όχι μόνο ε, τις αιμονές μας με την τεχνολογία και την έρευνα, αλλά να δούμε πώς μπορούν αυτά να εφαρμοστούν ε, εγκάρσια σε όλους τους κλάδους και βεβαίως με, με, τεχνικές ε, νέες για όλους. Για τις επόμενες γενιές θα πρέπει να τους δώσουμε τις δεξιότητες για να μπορέσουν να πετύχουν στη ζωή τους. Και κλείνω λέγοντας πως θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και την ηθική σχέση μεταξύ ε, όλων των επιπέδων της μικρής κοινότητας, της, ε, του έθνους, της ε, κοινότητας, του υπερεθνικού και να επενδύσουμε σε όλα αυτά τα επίπεδα στην παιδεία. Και πιστεύω πως θα τα καταφέρουμε, θα πετύχουμε όλοι μαζί ε, και θα κερδίσουμε όλοι και δεν θα καταλήξουμε σε μια εχθρότητα μεταξύ των εχόντων και των μη εχόντων. Θα πρέπει λοιπόν αυτά τα σχέδια να δημιουργήσουν μια νέα οικονομία ψηφιακή, ανοιχτή σε όλους, που θα έχει ωφέλη και θα εκτήματα για όλους εμάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα τώρα να συνεχίσουμε με την κυρία Ρωσία Δεφρούτος από την Ισπανική Βουλή. Καλησπέρα σας. Είμαι πολύ ευχαριστημένη που είμαι εδώ σήμερα γιατί το θέμα μας αφορά ιδιαίτερα και το κόμμα μου πιστεύει πως η ψηφιακή οικονομία, η ρομποτική, οι ψηφιακές πλατφόρμες, τα δίκτυα βάζουν μεγάλα στοιχεία καινοτομία στις εργασιακές σχέσεις και τις αλλάζουν από αυτό το σχήμα που γνωρίζουμε σήμερα. Βεβαίω υπάρχουν πολλές αμφιβολίες, δηλαδή πόσες θέσεις εργασίας θα χαθούν, για παράδειγμα, πώς θα δημιουργηθούν, τι δεξιότητες θα χρειαστούμε. Εγώ θα προσπαθήσω να απαντήσω σε τρία ερωτήματα που για τη δική μου ομάδα είναι πολύ σημαντικές και που βλέπουν το θέμα της ψηφιοποίησης από την ανθρώπινη πλευριά με σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Και γιατί, γιατί ανησυχούμε. Θα ξεκινήσω με ένα θέμα το οποίο είναι ζωτική σημασία για μένα. Ψηφιοποίηση. Η ψηφιακή οικονομία καταφθάνει σε μια συγκεκριμένη στιγμή όπου στις εργασιακές ε, σχέσεις αυτή τη στιγμή πρετανεύει η αβεβαιότητα. Δηλαδή θα προσθεθεί σε εργασιακές σχέσεις που έχουν χειροτερεύσει, φτωχοποίηση εργαζομένων, μερική απασχόληση, ε, συμβασιούχοι με ε, βραχυπρόθεσμες συμβάσεις, δηλαδή είναι πολύ περίπλοκη όλη η κατάσταση, μεγάλη ανασφάλεια και λέω πράγματα τα οποία συμβαίνουν στη χώρα μου και σε αυτά ε, προσθέτουμε νέα στοιχεία που αυξάνουν την επιβεβαιότητα. Για παράδειγμα, ψηφιακές πλατφόρμες. Ναι, μας τις προωθούν ως έναν τρόπο δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Και δεν λέω πως δεν αποτελούν κάτι τέτοιο. Αλλά τουλάχιστον στη δική μου χώρα δεν χρησιμοποιούν για αξιοπρεπή εργασία. Οι πλατφόρμες αυτές οι ψηφιακές στη χώρα μου τι δημιουργούν, όπως καταγγέλνουν τα συνδικάτα, νέους τρόπους εκμετάλλευσης. Και στην Ισπανία τουλάχιστον ουσιαστικά είναι και ο τελευταίος κρίκος στην αλυσίδα του φτωχοποιημένου εργαζόμενου. Γιατί έχουμε ένα νέο φαινόμενο. Η πλατφόρμα η ψηφιακή από μόνη της δεν είναι εργοδότης, δεν έχει συνείδηση. Οπότε όλοι οι εργαζόμενοι, για παράδειγμα, οι οδηγοί ε, που έχουν μηχανάκια ε, και δουλεύουν για κάποια τέτοια πλατφόρμα ουσιαστικά θεωρούνται ελεύθεροι επαγγελματίες χωρίς δικαιώματα. Ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι δεν το έχουν επιλέξει ως εναλλακτική λύση έτσι όπως μας πουλάνε αυτές οι ψηφιακές πλατφόρμες. Αυτό που συμβαίνει είναι, είναι εργαζόμενοι οι οποίοι το κάνουν γιατί δεν έχουν άλλη ευκαιρία δεν έχουν καμία άλλη δυνατότητα για να κερδίσουν το ψωμί τους. Και γι' αυτό κάνουν αυτή τη δουλειά. Και του συμπεριφερόμαστε σαν να είναι επαγγελμα... Ε, ελεύθεροι επαγγελματίε. Είναι αυτό το οποίο θα ε, ονομάζαμε στα ελληνικά μπλοκάκια με ένα μόνο εργοδότη. Οπότε καταλαβαίνετε τι προβλήματα δημιουργεί όλο αυτό και θα πρέπει να σταθούμε και να δούμε τι συμβαίνει μέσα σε ένα πλαίσιο όπου ουσιαστικά η αβεβαιότητα της απασχόλησης ουσιαστικά παγιώνεται μέσω αυτών των τεχνολογικών δυνατοτήτων. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε η ψηφιοποίηση να γίνει ένα ακόμα σκαλί ε, ε, που οδηγεί στην αυξημένη βεβαιότητα. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε τα δίκτυα αυτά να προσφέρουν θέσεις εργασίας που δεν είναι αξιοπρεπείς. Και υπάρχει και κάτι ακόμα που μας ανησυχεί. Προφανώς, και εδώ θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Θα μιλήσω για δίκτυα. Είμαστε, δια... Είμαστε δικτυωμένοι, υπερενημερωμένοι, υπερεκτεθειμένοι σε υπερσυνδέσεις και αυτό μας βοηθάει βέβαια να διαχειριστούμε τους ανθρώπινους πόρους, έχει κάποια πλεονεκτήματα, αλλά μην ξεχνάμε πως ουσιαστικά οδηγούμαστε σε καταστάσεις οποίες δεν γνωρίζαμε στο παρελθόν με τα εργασιακά δικαιώματα και να αναγνωρίσουμε πως όλα αυτά τα θέματα μπορεί να οδηγήσουν σε καταστάσεις ε, ακραίας ανασφάλειας για τους εργαζομένους που μπορεί να επηρεάσουν τη ιδιωτική του ζωή, για παράδειγμα στις ώρες εργασίας. Θα πρέπει να είναι μονίμως διασυνδεδεμένη και στην υπηρεσία της επιχείρησης. Μπορεί να επηρεάσει και τον κίνδυνο στον οποίο εκτίθεται κάποιος εργαζόμενος. Γιατί έχουμε αυτή την υπερέκθεση η οποία μπορεί να είναι επικίνδυνη. Και όλα αυτά θα πρέπει τα κράτη να τα τοποθετήσουν στα πλαίσια ενός νέου εργασιακού δικαίου που θα ισχύει σε κάποιες περιπτώσεις ε, ίσως περισσότερο, ίσως λιγότερο, γιατί αυτή τη στιγμή τα εργασιακά παντού καταραίων. αλλά θα πρέπει τουλάχιστον να έχουμε στο νου μας. Και τρίτον, η κατάρτιση, η εκπαίδευση, η επιμόρφωση είναι ζωτική σημασία για όλους, κυρίως όταν αναφερόμαστε στην ψηφοποίηση. Αλλά τι συμβαίνει. Στην πραγματικότητα η ανάγκη κατάρτισης κρύβει και μια μικρή παγίδα. Γιατί από την Ισπανία που είμαι εγώ, πάνε πολλοί πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε την ε, επιταγή, το βάτσο για την νεολαία κτλ. Αλλά δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να εκπαιδεύσουμε τους νέους μας για το αυτό που έρχεται. Όχι, τους έχουμε εκπαιδεύσει για κλάδους οι οποίοι ήδη έχουν πολύ ψηλά επίπεδα βεβαιότητας, για παράδειγμα έχουν αυτές τις ε, εργασιακές συμβάσεις ε, που επιδοτούνται. Γιατί? Για να ε, δουλέψουν στον χώρο της εστίασης, για παράδειγμα, ως καυσόνια. Δεν νομίζω ότι αυτό τους δίνει ιδιαίτερα προσόντα για τον ψηφιακό κόσμο και είναι κάτι το οποίο με ανησυχεί ιδιαίτερα. Υπάρχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι οι οποίοι, τους οποίους θα διώξουν θα τους πετάξει έξω η αγορά εργασίας και δεν θα μπορέσουν να ξανανεύουν στο τρένο ποτέ, γιατί δεν θα έχουν καταρτιστεί κατάλληλα. Για παράδειγμα, για όσους είναι πάνω από τα 50. Αν δεν θέλουμε να ζήσουμε λοιπόν σε μια κοινωνία αποξενωμένη, διαστροφική, ασθενή, θα πρέπει να τα προσέξουμε όλα αυτά, γιατί όλοι αυτοί θα μείνουν εκτός και δεν θα μπορέσουν ποτέ να ξανανεύουν επάνω στο τρένο. Θα έχουν κλείσει οι πόρτες της αγοράς εργασίας και είναι πολύ δύσκολο να φανταστώ πώς θα καταφέρουν να τις ξανανοίξουν. Και δεν θα μπορούν να δουλέψουν σε ένα ψηφιακό κόσμο. Αυτά είχα να σας πω. Είναι αλήθεια πως η ψηφιακή οικονομία θα μας δώσει πολλές δυνατότητες. Είναι αλήθεια πως υπάρχει και δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε καθόλου αυτό απλώς να είναι ένα ακόμα σκαλεί προς την αβεβαιότητα και ήδη η εργασία έχει γίνει πάρα πολύ αβέβαιη και οι, οι κοινωνικοί εταίροι και τα συνδικάτα έχουν χάσει μεγάλο κομμάτι της ισχύω τους. Η στιγμή είναι δύσκολη, περίπλοκη και πιστεύω ότι δεν θα πρέπει επουδενή να επιτρέψουμε η ψηφιοποίηση, η ρομποτική, τα δίκτυα, οι πλατφόρμες να μας οδηγήσουν σε πιο φτωχούς εργαζομένους και σε πιο πολλούς εργαζομένους οι οποίοι δεν μπορούν πια να απολαμβάνουν μια αξιοπρεπή εργασία. Σας ευχαριστούμε. Α, κύριε φρούτος. Δίνω τώρα το λόγο στην κυρία Κλάουδια Μούλερ, βουλευτή της α, ε, Γερμανικής ε, Βουλής. Ευχαριστώ. Δεν θα επαναλάβω τα όσα υπόθηκαν ήδη από του προηγούμενου ομιλητέ, απλώ θα τονίσω κάποια ακόμα στοιχεία συμπληρωματικά. Γνωρίζουμε πω η ψηφιοποίηση αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα σημεία καμπή ε, από τη βιομηχανική επανάσταση. Και αυτό σημαίνει ότι κάποιε θέσει εργασία ή κάποιοι τομεί θα εξαφανιστούν, αλλά θα προκύψουν νέοι τομεί εργασία. Η βαρέες εργασίες θα αντικατασταθούν στο μέλλον όλο ένα και περισσότερο από ρομπότ και από μηχανήματα. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι οι άνθρωποι θα μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα ε, στις ε, εργασίες τους και καθώς ε, και εμεί εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και άλλα σημεία στον κόσμο πλήττονται από τη δημογραφική αλλαγή, σημαίνει αυτό ότι θα πρέπει να προσαρμοστούμε καλύτερα στα όσα έχουμε μπροστά μας. Ε, καταρχήν, ε, υπάρχει ε, το ζήτημα της, του υψηλότερου προσδόκιμου ζωής. Αυτό αποτελεί μια πρόκληση, αλλά και κάτι το θετικό, γιατί βέβαια σημαίνει ότι διάφοροι εργαζόμενοι θα μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους στις επιχειρήσεις τους και αυτό σημαίνει με τη σειρά του ότι θα πρέπει να δούμε πώς οι εργαζόμενοι θα μπορούν να ελοποιήσουν καλύτερα ε, την, ε, το σκεπτικό και τη συλλογιστική της διαβίου μάθησης όχι μόνο όταν βρίσκονται σε κατάσταση ανεργίας αλλά και σε όλη τη διάρκεια του εργασιακού τους ε, βίου. Και αυτό βέβαια δεν αφορά μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες υποεκπροσωπούνται στη Γερμανία σε ό,τι αφορά ειδικότερα ακριβώς την παροχή ευκαιριών περαιτέρω επαγγελματική κατάρτισης. Από εκεί και μετά η δημιουργία ενός πιο δημιουργία ενό πιο συμμετοχικού χωρίς αποκλεισμούς ε, τομέα εργασίας συνδέεται ακριβώς με αυτή την ψηφιοποίηση. Δηλαδή η ψηφιοποίηση μπορεί να οδηγήσει στην καλύτερη προσβασιμότητα στην αγορά εργασίας μέσω τεχνικής υποστήριξης και κατά συνέπεια ε, καλύτερη ένταξη εργαζόμενων στην ε, αγορά εργασίας. Εδώ λοιπόν δημιουργεί πραγματικές ευκαιρίες η ψηφιοποίηση. Μία από τις βασικές προϋποθέσεις για να επιτευχθεί αυτό και στο οποίο δεν έχουμε επιτύχει ακόμα ε, το, αυτά όσα θέλουμε και στη Γερμανία είναι η τεχνική υποδομή. Δηλαδή για να το επιτύχουμε αυτό, να μεταλλευτούμε αυτές τις ε, ευκαιρίες ε, της ψηφιοποίησης θα πρέπει να έχουμε την κατάλληλη τεχνική υποδομή και μάλιστα σε όλες τις περιοχές. Αλλιώ θα επαναληφθεί η κατάσταση που είχαμε δει για παράδειγμα στον 19ο και τον 20ο αιώνα όπου για παράδειγμα κάποιες περιοχές οι οποίες ήταν ιδιαίτερα εύπορες και κάποιες ε, που βρίσκονταν ε, σε πολύ χειρότερη ε, κατάσταση. Και σήμερα, για παράδειγμα, βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές στην Γερμανία όπου η μέση ταχύτητα της σύνδεσης είναι γύρω στα 10 Mbit. Από εκεί και μετά. Η ψηφιοποίηση μπορεί να δημιουργήσει περισσότερε δυνατότητε home office, αλλά και καλύτερη, ε, καλύτερο συνδυασμό επαγγελματική και οικογενειακή ε, ζωή. Ταυτόχρονα όμω ε, σημαίνει ότι θα πρέπει να μεταβάλουμε τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων. Δηλαδή θα πρέπει να προσαρμοστούν τα όσα αδιέπουν του χρόνου ανάπαυση, του χρόνου ταξιδίου. Γιατί εάν δεν λάβουμε υπόψη μα και αυτέ τι διατάξει, ουσιαστικά θα επιτύχουμε το αντίθετο από αυτό που θέλουμε Δηλαδή, αντί να επιτύχουμε καλύτερη, ε, ε, καλύτερο συμβασμό μεταξύ επαγγελματική και οικογενειακή ζωή, τελικά θα δημιουργήσουμε μεγαλύτερε αντιθέσει μεταξύ του. Άρα, λοιπόν, θέλουμε να συνοδευτούν οι νέε δυνατότητε που δίνονται για του εργαζόμενου από υψηλότερο επίπεδο προστασίας των εργαζομένων. Κάτι ακόμα που θα ήθελα να αναφέρω είναι ε, κάτι που αναφέρθηκε έτσι συντομία, είναι αυτοαπασχολούμενο. Από το 2012 στη Γερμανία βλέπουμε ότι υπάρχει μια σημαντική αύξηση του ποστού αυτοαπασχολούμενο και θεωρούμε πως ε, ε, κάποιες νέες πλατφόρμες οι οποίες θα δημιουργηθούν ε, θα ε, ουσιαστικά καταστήσουν λίγο πιο ασαφή τα όρια μεταξύ της μισθωτής εργασίας και της ανεξάρτητης εργασίας. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να επιτύχουμε για παράδειγμα και κάποιες προστασίες τύπου ελάχιστου εισοδήματος και στον τομέα των αυτοαπασχολούμενων έτσι ώστε να αποφύγουμε φαινόμενα κοινωνικού dumping. Κάτι τέτοιο δηλαδή θα πρέπει να το διασφαλίσουμε βλέποντας και πώς μπορούμε να συμμορφωθούμε με τα όσα βλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία νομοθεσία και το αναφέρουμε ειδικότερα και στην τελευταία οδηγία σε ό,τι αφορά την παροχή υπηρεσιών. Θα πρέπει, για παράδειγμα, να δούμε πώ οι νέε μορφέ εργασία θα περιληφθούν και στα συστήματα κοινωνική ασφάλιση και θα πρέπει να δούμε πώ μπορούμε να συμπεριλάβουμε σε όλο αυτό το νέο σύστημα και τι πολύ μικρού μεγέθου επιχειρήσει. Είναι ζητήματα τα οποία απασχολούν αυτή την περίοδο τη δική μα ε, ε, χώρα ε, και η δική μας Υπουργό Εργασίας είχε υποβάλει μια λευκή βίβλο με 177 σελίδες ε, όπου όμως δεν αναφέρονται συγκεκριμένες λύσεις. Συγκεκριμένες λύσεις τις οποίες δηλαδή θα πρέπει τώρα εμείς να καταρτήσουμε, να συντάξουμε να σκεφτούμε μέσα στα επόμενα χρόνια. Και βέβαια πάντοτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί τέτοιου είδου λύσει μόνο ευρωπαϊκό προσανατολισμό μπορούν να έχουν και γι' αυτό το λόγο χαίρομαι και τη συζήτηση που κάνουμε σήμερα εδώ μεταξύ μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ε, την κυρία Μίλλερ. Κλείνοντας ε, θα ήθελα να δώσω και πάλι το λόγο στον κύριο Γιώργη Γιώκοφ ο οποίο είναι ο επικεφαλή ε, τη Κοινοβουλευτική Επιτροπή για Συστήματα Εργασία ε, τη Εθνοσυνέλευση τη Βουλγαρία. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αποτελεί χαρά μου το να βρίσκομαι σήμερα εδώ για να συζητήσουμε κάποια ζητήματα τα οποία μας απασχολούν όλους μας γιατί πράγματι το μέλλον της ψηφιοποίησης αποτελεί σημαντικό ζήτημα για, όλα, για όλες τις χώρες. Στο παρελθόν η βιομηχανική επανάσταση είχε ένα μεγάλο βάθος χρόνου, ενώ αντιθέτως οι αλλαγές τις οποίες βλέπουμε τώρα ε, λαμβάνουν χώρα μέσα σε δεκαετίες. οι πρώτε, ε, για παράδειγμα, αλλαγέ ξεκίνησαν ακριβώ πριν από μερικέ ε, δεκαετίε. Η ψηφιοποίηση λοιπόν πολύ γρήγορα επιβλήθηκε και ε, αποτέλεσε βασικό κομμάτι όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων. Ε, η ίδια δηλαδή παραγωγικότητα ε, μπορεί πλέον να επιτευχθεί ε, με 50-70% λιγότερο εργατικό δυναμικό από ό,τι αυτό συνέβαινε στο παρελθόν και αυτό ισχύει και στου τομεί της μεταποίηση και στον τομέα των ε, γεωργικών. Δηλαδή ε, βλέπουμε πόσο ε, σημαντικό ρόλο παίζει εδώ η ψηφιοποίηση. Η ταχύτητα μάλιστα με την οποία συμβαίνουν όλα αυτά αφορά όχι μόνο τον οικονομικό τομέα αλλά γενικότερα τον κοινωνικό τομέα και βλέπουμε ότι υπάρχουν ολοένα και περισσότερε προποθέσει, οι οποίε ισχύουν σε ό,τι αφορά τον τομέα τη παιδεία και τη κατάρτιση. και βρισκόμαστε ουσιαστικά δηλαδή εν μέσω μιας τέταρτης ε, επανάστασης ε, ε, στο πλαίσιο της οποίας οι εργαζόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν νέες, νέα επαγγελματικά προσόντα, νέες δεξιότητες. Βέβαια είναι ακόμα νωρίς για να πούμε από τώρα πού θα μας οδηγήσουν όλες αυτές οι αλλαγές, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που είναι αδιαφυσβήτητο είναι ότι η τεχνολογία μεταλλάσσεται ταχύτερα από ό,τι οι νοοτροπίες και συνήθειες των εργαζομένων. Ουσιαστικά δύο ρεύματα σκέψης υπάρχουν σε ό,τι αφορά αυτή την ψηφιοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη μία πλευρά δηλαδή ε, θεωρείται ότι μπορεί να, υπάρξει, ε, να υπάρξουν ε, περισσότερες κοινωνικές ανισότητες ενώ κάποιοι πιστεύουν ότι ε, μπορεί να υπάρξει και συρρήκνωση της ε, ε, οικονομίας κατά 40-50% στο 2050. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ένα ρεύμα σκέψη, το οποίο είναι πιο αισιόδοξο και θεωρεί ότι ουσιαστικά ε, δημιουργούνται νέοι ορίζοντες, νέες ευκαιρίες, αφού θα έχουμε πιο εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό ε, και εργασιακές ευκαιρίες οι οποίες θα εστιάζουν ιδιαίτερα ε, στην καινοτομία και στην δημιουργικότητα. Καθώς και η τα σύνορα, τα όρια, αν θέλετε, τα εμπόδια σε ό,τι αφορά την αγορά εργασία και την παραγωγή θα, δεν θα υπάρχουν πλέον. Αν πάντως ε, θέλουμε να κινηθούμε εδώ ως ε, σύνολο στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιτύχουμε περισσότερη σύγκληση μεταξύ μας. Θα πρέπει λοιπόν οι προσπάθειες που κάνουμε εδώ να εντάσσονται σε ένα γενικότερο πλαίσιο για να μην επιτρέψουμε ε, την δημιουργία ή την ύπαρξη μιας Ευρώπης δύο ταχυτήτων. Η ψηφιοποίηση επηρεάζει τη ζωή των ανθρώπων και σίγουρα θα μεταβάλει δράστικα την αγορά εργασίας. Εάν λοιπόν χάθηκε το 40% ε, των θέσεων εργασίας λόγω ακριβώς ε, της ε, εκβιομηχάνησης της παραγωγής. Τώρα αναμένουμε λόγω της ψηφιοποίησης να χαθεί ένα συμπληρωματικό 10-15% των θέσεων εργασίας. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η απώλεια των θέσεων εργασίας. Και ενώ έχει γίνει μια συζήτηση σε επίπεδο ενός ακόμα, υπάρχουν διάφορες ε, στις Για παράδειγμα, τα δικαιώματα των εργαζομένων ε, και οι σχέσεις ε, των κοινωνικών εταίρων είναι σημαντικά. Δηλαδή, η ψηφιοποίηση θα επηρεάσει τις σχέσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων καθώς και η συλλογική διαπραγμάτευση και Ε, το 2020 η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει 25 ε, εκατομμύρια ενέργους. Ε, πώς λοιπόν θα βρούμε τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι θα είναι σε θέση να καλύψουν τις σχετικές θέσεις εργασίας. Ουσιαστικά αυτό που χρειαζόμαστε είναι άνθρωποι με τις κατάλληλες αποτελεσματικές δεξιότητες, τα κατάλληλα προσόντα. Οπότε θα πρέπει να αξιοποιήσουμε όλο το δυνατό δυναμικό που έχουμε στη διάθεσή μας, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τους εκπαιδευτές, ε, την κοινωνία των πολιτών, όλους λοιπόν όσοι μπορούν, ε, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε από κοινό τις ε, προκλήσεις αυτές. οι πολίτες δηλαδή θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλαμβάνουν δραστηριότητα και ω επιχειρηματίε ε, στον χώρο τη και με αυτόν τον τρόπο να δημιουργούν με τη σειρά του νέε θέσει εργασία. Οι καινοτόμε τεχνολογίε ε, και η δημογραφική αλλαγή ε, καθιστούν απαραίτητε κάποιε νομοθετικέ τροποποιήσει. Τροποποιήσεις βέβαια τις οποίες θα πρέπει να κάνουμε μετά από μια προσεκτική ανάλυση τη κατάσταση. Χρειαζόμαστε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο θα διασφαλίζει ε, την ισότητα, την ε, οικονομική ανάπτυξη αλλά και θα ε, προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων. Η ψηφιοποίηση ουσιαστικά δημιουργεί ένα νέο μοντέλο, καταργεί το, ε, μέχρι το, το υφιστάμενο ε, μοντέλο εργασίας, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί και αλλαγές σε ό,τι αφορά τον τρόπο ζωής των ανθρώπων. Ουσιαστικά ε, ο επαγγελματικό βίος γίνεται όλο και πιο μεγάλος, δηλαδή καταλαμβάνει περισσότερες ώρες της ημέρας και Εμείς ε, ε, στην ε, Βουλγαρία έχουμε, προετοιμάζουμε μία σειρά από μέτρα σε ό,τι αφορά αυτή την τέταρτη επανάσταση ακριβώς λόγω και της δημοκρατικής αλλαγής και των νέων αναγκών οι οποίες θα προκύψουν με πάση την νέα κατάσταση. Ε, κλείνοντας να πω ότι εάν ρίξουμε μια ματιά στην ιστορία μας ε, θα διαπιστώσουμε ότι η φόβη μας σε ό,τι αφορά την ψηφιοποίηση της ε, αγοράς εργασίας είναι μεν βάσιμε, αλλά από την άλλη πλευρά θα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Δηλαδή, σε τελική ανάλυση τελικά μπορεί να αποδειχθούν ε, ω ε, αβάσιμε και γι' αυτό αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τη συζήτηση η οποία θα γίνει στο επίπεδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τα συμπεράσματα από αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Γιώκοφ. Να σα θυμίσω ότι ο χρόνο ε, ομιλία είναι περιορισμένο. Έτσι θα μπορούν να μιλήσουν περισσότεροι. Δύο λεπτά είναι το όριο. Μετά λοιπόν από τις διάφορες εισαγωγικέ δηλώσεις να δώσω το λόγο στον πρώτο που ζήτησε το λόγο. Την κυρία Μαρία Σκου. έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ήθελα να πω ότι κατά διάρκεια αυτής της θητείας, η Ιταλικής θητείας στο Κοινοβούλιο, που ολοκληρώνεται η θητεία του Ιταλικού Κοινοβουλίου, μελετήσαμε τον αντίκτυπο των εκλογικών εξελίξεων όσον αφορά την αγορά εργασία και την οικονομία. Δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή και προβληματισμό πάνω σε αυτό οι δύο οι επιτροπές, οι διάφορες αρμόδιες του Κοινοβουλίου επεξεργάστηκαν μια έρευνα, κάναν μια έρευνα που οδήγησε στην έγκριση ενός εγγράφου με συμπεράσματα που αναφέρθηκε σε προβληματισμούς που αφορούσαν τις επιχειρήσεις, πώς μπορούν να απτυχθούν μέσω ψηφιακών εξελίξεων και πώς μπορούν να ανταγωνιστικές του το τρόπο σε παγκόσμιο επίπεδο και πώς θα προστατευθούν οι περιφέρειες και οι πολίτες οι πιο ευάλωτοι από αυτή τη μεταμόρφωση τη βιομηχανική. Διαφάνει λοιπόν ότι κάποιες θέσεις απασχόλησης σίγουρα θα απολεστούν και κάποια επαγγέλματα μόνο εν μέρη θα μπορέσουν να, αλλά, να προσαρμοστούν. Αυξάνεται η ζήτηση κάποιες δεξιότητες. Άρα χρειάζεται επέκταση και διάδοση διαφόρων τρόπων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στην Ιταλία αυτά τα προβλήματα γίνονται ιδιαίτερα αισθητά, διότι το ποσοστό των εργαζομένων που απασχολούνται στην βιομηχανία ε, είναι το, από, τα, από τα υψηλότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε επιβεβαιώνεται εκεί η τάση που διαπιστώνει σε διεθνέ επίπεδο. Σε εμά όμως, στην Ιταλία, οι ανισότητες σίγουρα θα είναι μεγαλύτερες. Για αυτού του λόγου θεωρούμε απαραίτητο να παρέμβουμε όσον αφορά την παιδεία και την κατάρτιση, επαγγελματικό προσανατολισμό, σε αυτούς τους τομείς να παρέμβουμε. Να σας πω λοιπόν ότι όσον αφορά την πτυχή της κατάρτισης, πρόσφατα, πειραματικά, στην Ομοθεσία του υπολογισμού του 2018, θεσπίσαμε για ένα χρόνο ε, μία πίστοση για τους εργοδότες, πειραματικά, στην Ομοθεσία του του 2018, θεσπίσαμε για ένα χρόνο ε, μια πίστοση για τους εργοδότες τα βάση διαφόρων προγραμμάτων το προγράμματος 4 κατάρτισης. Περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ δίδονται για αυτούς τους όρους. Τίθενται όροι μέσω συλλογικών συμβάσεων ή περιφερειακών ε, συμβάσεων όσον αφορά την εφαρμογή αυτού του προγράμματος ε, κατάρτισης των εργαζομένων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Σβετλάνα Αγγέλοβα της Επιτροπής Εργασίας τη της Εθνοσυνελεύσεως της Βουλγαρίας στο χώρο εργασίας και στην αγορά εργασίας και στη ζήτηση για διάφορου διάφορους εργαζομένους με δεξιότητες. Δυναμικές οι αλλαγές που συνεπάγονται τάσεις παρόλο που σε κάποιους τομείς οικονομίας οι εξελίξεις είναι πολύ ταχύτερες και πολύ πιο έντονες. Ε, η ψηφιοποίηση δική εργασία, επίλυση προβλημάτων. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να δράσουν έγκαιρα, ούτως ώστε να εξασφαλίσουν το τομέα της ψυχικής τεχνολογίας. Το να καθορίζουμε τα σωστά προσόντα που ψάχνουν οι εργοδότες προσφοράς και ζητήσεως στην αγορά εργασίας είναι αναπόσπαστο κομμάτι Τη παραγωγική απασχόληση υψηλή ποιότητα. Έτσι θα εξασφαλίσει μέτρα και νομοθεσία ώστε να εξασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο προστασία για το εργατικό δυναμικό συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων, Οι οποίοι αυτοαπασχολούμενοι πολύ συχνά ηγούνται στη νέα τεχνολογία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Αγγελόβα. Και τώρα ο κύριος Νικόλας Μάνιος, ε, που είναι πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Συνάδελφοι και συνάδελφοι και συναδέλφισες, ε, χαίρομαι που είμαι πάλι μαζί σας να συζητήσουμε ένα πολύ κρίσιμο θέμα. Έχουν εμφανιτέλημα ο εργαζόμενος να μην προστατεύεται από το εργατικό δίκαιο η Ελλάδα προέκρινε μια σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν τι ευέλικτε μορφέ απασχόληση, άτυπε μορφέ απασχόληση, στην παροχή αποτελεσματικών εγγυήσεων, όπου οι φυστάμενε ρυθμίσει δεν επέτρεψαν τη δημιουργία να μην επιτρέψουν λόγω του είδου τη σχέση τη σύμβαση εργασία. Είναι φανερό ότι η ψηφιοποίηση τη εργασία απαιτεί εξειδικευμένε ψηφιακέ γνώσει, κάτι που είναι πρώτη στο καθήκον για τις μέλη και για τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να προχωρήσουν σε μια επέκταση της δυνατότητας απόκτησης αυτών των ε, ψηφιακών νέων γνώσεων και δεξιοτήτων. Πρέπει να λειτουργεί επέκταση της δυνατότητας απόκτησης αυτών των ε, ψηφιακών νέων γνώσεων και δεξιοτήτων. Πρέπει να λειτουργικότερης κρίσης και ανισότητας θα αναφερθώ αναγκαστικά για το χρόνο της ελάχιστος στη φράση που είπε ο Πρωταγόρας χιλιάδες να συμβάλλει και να τα λύσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Γιον Κυρίους που είναι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε συνάδελφοι για να συζητήσουμε ένα θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο είναι ότι έθεσε το μέλλον της εργασίας στην ημερήσια διάταξη. Και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εργασίας ασχολείται με το θέμα αυτό και έχουμε συναδέλφους οι οποίοι εργάζονται σκληρά για να δούμε ποιο θα είναι το μέλλον της εργασίας, για να προοδεύσουμε σε όσα κάνουμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το μέλλον. Και θα ήθελα να σταθώ στα σχόλια που έγιναν από όσους δουλεύουν για ψηφιακές πλατφόρμες βλέπετε πως αυτές οι εταιρείες που βασίζονται σε πλατφόρμες συνήθως που βρίσκονται σε περισσότερο από ένα κράτη-μέλη, αλλά υπάρχουν σε πολλά κράτη-μέλη και που προσπαθούν να προωθήσουν τις πολιτικές τους. αναρωτιόμαστε πώς μπορούμε να κάνουμε πιο ευέλικτη την αγορά εργασίας. Όταν λοιπόν το συζητάμε θα πρέπει να σκεφτόμαστε τι είδους Action. Όταν μεταρρυθμίζουμε την αγορά εργασίας θα πρέπει να απλουστεύουμε το εργασιακό δίκαιο, να εξασφαλίζουμε όταν μεταρρυθμίζουμε την αγορά εργασία, θα πρέπει να απλουστεύουμε το εργασιακό δίκαιο, να εξασφαλίζουμε πως ο κόσμος θα μπορεί μέσα σε αγορά εργασίας να προοδεύσει και να προχωρήσει και αυτό πως προσφέροντας μια σφαιρική ποιότητά τους και θα μειώσει τον κίνδυνο της ανεργίας. Επίσης η γύρανση του εργατικού μας δυναμικού και αυτό είναι μια πρόκληση και χρειάζεται μέσα στη... Ε, δηλαδή μέτρα τα οποία θα αυξήσουν τα επίπεδα ευαισθητοποίησης για το θέμα αυτό όπου οι επιχειρήσεις θα γνωρίζουν καλύτερα σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο. Oh, Σας ευχαριστώ πολύ. Θεωρήσουμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα περιβάλλον ελκυστικό για την ψηφιακή οικονομία, για την οικονομία υψηλής τεχνολογίας, για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλο το δυναμικό της ψηφιακής οικονομίας. Μετά θα μπορούσαμε να δούμε και ποια θα είναι η κοινωνική ομπρέλα προστασίας και τα δίκτυα, σίγουρα θα χαθούν πολλές θέσεις εργασίας. Αυτό είναι βέβαιο. Ή θα αναδιαστρωθούν. Είχαμε και μία μελέτη για εννέα βόρειες χώρες, πολύ πρόσφατα δημοσιεύθηκε από την Μακέντζη και την ψηφιακή οικονομία με φόβο. Θα πρέπει απλώς να εξασφαλίσουμε πως το περιβάλλον και το επιχειρηματικό περιβάλλον ε, θα προσελκύσει τις νέες ευκαιρίες και πως θα έχουμε περισσότερες θέσεις εργασίας και κοινωνική ομπρέλα προστασίας που είναι αυτό το οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στη Σοφία Ριμπέιρο. Ευχαριστώ πολύ κύριε ε, την ε, ρομποτική και το ότι αποτελούν όλες αυτές τις πτυχές μέρος μιας νέας ανάπτυξης, μιας νέας εξέλιξης, η οποία ήδη έχει ξεκινήσει. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα σε έναν κόσμο ή δύο όπου το να μπορεί κανείς να προγραμματίζει τον υπολογισμό, ε, στον υπολογιστή συγγνώμη, είναι τόσο σημαντικό όσο και το να ε, γράφει και να διαβάζει. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προετοιμάσουμε και τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας έτσι ώστε να είναι έτοιμες για να αντιμετωπίσουν αυτές τις νέες προκλήσεις. Θα πρέπει να τελειώσουμε τους ε, νέους μας αλλά και τους καθηγητές ούτως ώστε να μπορέσουν να συμβάλλουν στην κατάλληλη εκπαίδευση των νέων. Θα πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε ταυτόχρονα και στην διαβιομάθηση έτσι ώστε να μπορέσουμε να συντονίσουμε καλύτερα και τις γνώσεις τις οποίες παρέχουν τα ακαδημαϊκά μας ιδρύματα ε, στα όσα είναι απαραίτητα ε, για τις επιχειρήσεις στον τομέα της ε, ρομποτικής και της ιοντομίας. Κάτι ακόμα τώρα με το οποίο θα πρέπει, το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι το να ακριβώς να προσαρμοστούμε χωρίς όμως να υπάρχουν, να υπάρχουν αυξήσεις των ανισοτήτων και περιφερειακών και κοινωνικών. Για παράδειγμα εγώ προέρχομαι από μια εξαιρετικά απόκεντρη περιοχή και ακριβώς προκύπτει αυτό το πρόβλημα, δηλαδή του πώς θα μπορέσουμε μπορέσουμε να δώσουμε τις καλύτερες γνώσεις στους αγρότες μας και όσα χρειάζονται αφού η κατάσταση η οποία ισχύει για τη δική μου περιοχή ισχύει για μία σειρά περαιτέρω περιοχέ τη ε, Πυρτουκή Πορτογαλία. Δηλαδή, πώ μπορούμε να ε, δώσουμε τι κατάλληλε ευκαιρίε ε, σε αυτέ τι περιοχέ, οι οποίε δεν είναι και κατοικημένε και στι οποίε δεν υπάρχει κατάλληλη πρόσβαση στην απαραίτητη κατάρτιση. Κάτι ακόμα, μία ακόμα πρόκληση είναι η προσαρμογή τη αγορά-εργασία αλλά και τη δημοσιονομική πολιτική, έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη οι νέε μορφέ εργασία. Εδώ αναφέρομαι ιδιαίτερα στην κινητικότητα στο πλαίσιο της εργασίας, αναφέρομαι ειδικότερα ε, στα μοντέλα ε, μέρικης εργασίας ή εξαποστάσεω εργασίας, τα οποία θα πρέπει να συμβάλλουν στην συμμετοχή, στην αύξηση συμμετοχή και όχι στον αποκλεισμό από την αγορά εργασία των ατόμων που διαβιούν ακριβώ σε πιο απομακρυσμένε περιοχέ. Άρα λοιπόν ε, θα ήθελα σε αυτό το πλαίσιο ε, να ρωτήσω και τους ε, ομιλητές μας εδώ το πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε το καλύτερο τρόπο αυτές τις τρεις βασικές προκλήσει. Σα ευχαριστώ. Η κυρία Λάουρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει το λόγο. Очевидно ναι. е, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ που αναφέρατε τις εμπειρίες σας, τις κοινοβουλευτικές που έχω. Από αυτά που βλέπω είναι ότι η πραγματικότητα ε, πρέπει να παρακολουθείτε και να συγχρονιστούμε με αυτή εμβάθυνση των ικανοτήτων, αλλαγή του συστήματος κατάρτιση είναι κάτι σημαντικό. Ενώ τα κάνουμε αυτά όμως για τους νέους μας που έχουν γίνει και να καταρτιστούν ξανά, να αποκτήσουν νέες απαιτούμενες δεξιότητες και σε θέσεις που καινούριου που απαιτούνται που είναι πολύ διαφορετικής νοημοσύνης της ρομποτικής. Να επενθυμίσω το Ευρωκοινοβούλιο τον περασμένο Οκτώβριο με μεγάλη πλειοψηφία υιοθέτησε το έγγραφό μας για το ελάχιστο και ε, είχα την εντύπωση από αυτά που άκουσα ότι όλα πάνε καλά. Όμως ε, πολύ σπάνια η πραγματικότητα τα αποκρίνεται στις μελέτες. Εδώ μιλάμε για ανθρώπινη διοργάνωση. Δεν υπάρχει καλή οργάνωση της αγοράς εργασίας όταν και ψηφιακή χωρίς να υπάρχει ανθρώπινη με το καφέ τους. Χρειάζεται αυτή η ανθρώπινη επαφή. Εγώ εργάστηκα στη Χαλιβουργία που ήταν πολύ ψηφιοποιημένη και κάθε φορά μα εξηγούσαν ότι θα μας διευκολύνει ψηφιοποίηση τη ζωή και κάθε φορά υπήρχαν τάσει διότι κάθε φορά λησμονούσαμε τι ανθρώπινε σχέσει, τι επαφέ. διότι είναι εργοστά, τα ρομπότ ε, μόνο του δεν κάνουν βρωμική εργασία αλλά και οι υπεργολαβίε δημιουργούν τα προβλήματα. Και πολύ συχνά αυτοί που αναλαμβάνουν τι υπεργολαβίε είναι άνθρωποι που πληρώνονται με πολύ χαμηλέ αμοιβέ και μετά τα πράγματα δεν είναι απλώς μηχανικά. Ίσως θα καταργηθούν θέσεις απασχολήσεως από ένα σημείο Β και θα δημιουργηθούν περισσότερες. Υπάρχει αυτή με την κατάσταση. Να το λάβουμε υπόψη. Όλοι, όλοι, όλοι δεν μπορούν να ασχολούνται με την πληροφορική, ούτε να είναι μηχανικοί. Τι θα κάνουμε στου υπόλοιπου. Ποιο είναι ο κίνδυνος, τι φοβάμαι. Θα δούμε ε, έναν κατακαιρματισμό της κοινωνική οικονομία. Θα έχουμε κοινωνίε που συγκατοικούν, αλλά δεν έχουν πολλά κοινά σημεία. Η οργάνωση σωστή αλλά και σε ανθρώπινο επίπεδο των φορέων των εργαζομένων και σωστή. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Ο κύριος Σούστερ, Ευρωβουλευτής, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Δεν μοιάζει να θέλει να πάρει το λόγο συνάδελφο. Ωραία λοιπόν, έκλεισε ο κατάλογος ομιλητών. Νομίζω ότι είναι προφανώ πως η συζήτηση αυτή για την ψηφιοποίηση και για το πώς θα επηρεάσει την αγορά εργασία, τις δεξιότητες, τα δικαιώματα, τι υποχρεώσει των εμπλεκομένων είναι θέματα τα οποία μας αγγίζουν πολύ βαθιά και τα οποία τώρα ξεκινάμε ε, να αντιμετωπίζουμε. Θα πρέπει λοιπόν να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και θα ήθελα τώρα να μου επιτρέψετε να καλέσω την Συμπρόεδρο ε, για να παρουσιάσει ε, το επόμενο κομμάτι της σημερινής συνεδρίας. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε λοιπόν στο δεύτερο τμήμα που αναφέρεται στις ανισότητες στα κράτη-μέλη. Έχουμε ήδη συζητήσει τις ανισότητες, αλλά τώρα μπορούμε να εστιάσουμε στο σημείο αυτό. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω να δώσετε το λόγο στον Ιβάν Μπαρτόλου, στον Γιάννη Κράινη, στη Ράκτα Μάξοβα και στην Σετλάνα Αγγέλοβα. Σας παρακαλώ πολύ, ελάτε συνάδελφοι να καθίσετε δίπλα μου. να μπούμε σε περισσότερο βάθος στο θέμα αυτό και θα ήθελα να ξεκινήσω με τον Ιβάν Μπάρτολο που είναι από τη Μάλτα, είναι μέλος του Κοινοβουλίου της Μάλτας. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή τη στιγμή διανύουμε μια εποχή της κοινωνικής και οικονομικής αλλαγής. Είναι σημαντικό λοιπόν για να έχουμε τάξεις στις κοινωνίες μας. Να είμαστε χαμηλά εισοδήματα και οι οικογένειες ζουν σε φτωχές ε, περιοχές. Τα παιδιά σε διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ενώ συμφωνούμε πως η κοινωνικονομική αλλαγή είναι σημαντική στη Μάλτα με υποπληροφορίες Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 70.000 άτομα κινδύνευσαν ε, 6. Είναι απαράδεκτο. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή ενισχύεται. Έχουμε τους καλύτερους ρυθμούς. Το 2016 είχαμε επίπεδα απασχόλησης παρόμοια με αυτά του 2008, δηλαδή της εποχής προκρίσης. Όμως, παιδείας είχαμε περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Είχαμε περισσότερες θέσεις στον κλάδο της επικοινωνίας, για παράδειγμα, σε πολλούς επιστημονικούς κλάδους. είχαμε τόσο γρήγορα, για παράδειγμα, στο χώρο της οικοδομής. Αλλά ναι, πολύ γρήγορα στις ενοικιάσεις. Και πρέπει να σας πω πως έχουμε και δωρά εργασίας στην Ευρώπη. Επίσης, στην ηλικία 45-65 η συμμετοχή των εργαζομένων ε, στην ε, κατά 2015 αυξήθηκε στη Μάλτα και τα άτομα μέχρι την ηλικία των 59 που κινδύνευσαν, ε, που βρίσκονται σε επίπεδα κοντά στο επίπεδο ξηθή οι κοινωνικές ασφαλίσεις που πληρώνουν οι εργαζόμενοι και έχουν μειωθεί οι συντάξεις που θα λάβουν όταν συνταξιδοτωθούν. Γιατί τα μελλοντικά συνταξιδοτικά συστήματα θα όσο δεν αντιστρέφουμε τις δημογραφικές τάσεις της χώρας μας και θα επηρεάσει όλους τους κλάδους που θα έχουν χαμηλότερα εργατικά δυναμικά. Okay, I'll try to stay below. θα προσπαθήσω να τηρήσω χρόνο μου. Αύριο είναι η μέρα της ε, κοινωνικής ε, δικαιοσύνης και της κοινωνικής ε, ισότητας, οπότε νομίζω πως είναι κατάλληλη χρονική συγκυρία για να αναφερθούμε στα ζητήματα ισότητας ή ανισότητας και παρατηρούμε πράγματι πως υπάρχουν διάφορες μόρφες ανισότητας μεταξύ των κρατών μελών μας σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τις ευκαιρίες, σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, σε ό,τι αφορά την κατανομή του εισοδήματος, σε ό,τι αφορά τον πλούτο, μια ανισότητα μάλιστα η οποία αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια ενώ <clears throat> ήδη είχαμε επιτύχει, ε, είχαμε επιτύχει αρκετή πρόοδο κατά τελευταία 100 χρόνια, αλλά και ανισότητα σε ό,τι αφορά το επίπεδο της εφορολόγησης, ε, για παράδειγμα. αν ε, κάνουμε μία σύγκριση ανάμεσα στα επίπεδα φορολόγησης των λιγότερων και των περισσότερων εφόρων, θα δούμε πως η φορολόγηση των εργαζομένων είναι πάντοτε ευξηνότερη. Ε, και επίση, ε, σε ό,τι αφορά το μέγεθο των επιχειρήσεων. Οι μικρέ επιχειρήσει καταβάλουν τελικά υψηλότερου φόρου ε, σε σύγκριση με μεγαλύτερε επιχειρήσει Οι μεγαλύτερε δηλαδή επιχειρήσεις όσο μεγαλύτερε είναι τόσο λιγότερου φόρου καταβάλουν. Έχουν δηλαδή τη δυνατότητα να αξιοποιούν προ όφελό τους την νομοθεσία οι μεγάλες επιχειρήσεις. Κάποιες τώρα από αυτές από αυτή τη διακριτική μεταχείριση ή μάλλον η ανισότητα την οποία παρατηρούμε βασίζεται ακριβώς στην ε, διακριτική μεταχείριση. Για παράδειγμα στο γεγονός ότι ε, γυναίκες ε, λαμβάνουν χαμηλότερα εισοδήματα σε σύγκριση με τους άντρες, κάποιοι οι οποίοι έχουν κάποια διαφορετική φυλετική καταγωγή, εθνοτική καταγωγή, έχουν λιγότερες ευκαιρίες απασχόλησης και από εκεί και μετά υπάρχει και ανισότητα σε ό,τι αφορά και τον νόμο, ενώπιον του νόμου. Και νομίζω καθώς ε, όλοι μας εδώ συμμετέχουμε στην νομοθετική διαδικασία, ε, θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε με τρία τίνα, τα οποία θα μπορούσαν να συμβάνουν στη μείωση αυτών των ανισοτήτων. Ένα από αυτά ε, αφορά την ανισότητα σε ό,τι αφορά την φορολόγηση. Αν δούμε για παράδειγμα το ακαθάριστο εισόδημα, δηλαδή ε, αυτή η πίτα αν θέλετε την οποία παράγει κάθε χώρα μας γύρω, το, ε, γύρω στο 60% ε, από αυτήν την πέτα το λαμβάνουν αυτοί οι, οι οποίοι εργάζονται, εργαζόμενοι και το υπόλοιπο 40% το οποίο εντάξει μπορεί να είναι λίγο υψηλότερο ή λίγο χαμηλότερο 30-50% το 40% αφορά ε, ε, τον, ε, τον, τους, τους φόρους από, αυτούς, από, την, από τον φυστόμενο πλούτο. Οπότε θα δούμε ότι σε ό,τι αφορά τους φόρους που αντιστοιχούν σε αυτή την πίτα, το 75% έως 90% και κατά κανόνα πάνω από το 80% είναι, προέρχεται από τους εργαζόμενους, οι οποίοι λαμβάνουν, όπως είπαμε, μόνο το 60% αυτής της ε, πίτας. Ενώ ε, όσοι λαμβάνουν το 40% αν θέλετε αυτής της πίτας, ε, μόνο καταβάλουν κατά 10 έως 15% φορολογικά σε αυτήν. Ε, και αυτό βέβαια βασίζεται στους νόμους τους οποίους εμείς έχουμε θεσπίσει. γιατί η φορολόγηση του κεφαλαίου έχει ένα συντελεστή της τάξης, του, της εργασίας έχει ένα ποσοστό, ένα συντελεστή της 40% ενώ η φορολόγηση του κεφαλαίου βρίσκεται γύρω στο 20%. Άρα λοιπόν η φορολόγηση έτσι όπως την έχουμε εμείς δημιουργήσει δημιουργεί περισσότερη ανισότητα. Εάν δούμε για παράδειγμα το πώς δημιουργούν τα αισθήματα της κληρονομίας, ε, κεφαλαϊκής ε, φορολόγησης, ε, μερισμάτων και ούτω καθεξής αφενός και φορολόγησης εργασίας αφετέρου, θα διαπιστώσουμε ότι η φορολόγηση της εργασίας είναι τουλάχιστον διπλάσια από ό,τι όλων των υπόλοιπων αυτό λοιπόν θα μπορούσε να μεταβληθεί και θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε περαιτέρω. Ε, τώρα, ένα δεύτερο ζήτημα είναι ε, το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο ανισότητα σε ό,τι αφορά την ε, κατανομή, η άνισο κατανομή του εισοδήματο. Ε, από ιστορική σκοπιά βέβαια υπήρχε αυτό και στο παρελθόν και υπήρξαν τρει μέθοδοι οι οποίε χρησιμοποιήθηκαν. Πρώτον οι επαναστάσει, δεύτερον μεγάλη, μεγάλη έκταση πόλεμη, οπότε βέβαια δεν θα ήθελα να προτείνω καμία από τι πρώτε δύο μεθόδου και τρίτης τρίτη μέθοδος ε, ήταν η προοδευτικού τύπου φορολογήσεις ε, ακριβώς ε, του ερυφαλού και της κληρονομίας και έτσι μέσα σε μερικές γενιές ήταν δυνατόν να υπάρξει καλύτερη κατανομή του εισοδήματο σε αυτές τις χώρες. Βέβαια, χωρίς να έχει λάβει χώρα κάποιος ε, πόλεμος ε, στην επικράτηση των ΗΠΑ. Ε, αν εξαιρέσουμε το Pearl Harbor, το οποίο δεν μπορούμε βέβαια να θεωρήσουμε ότι είχε κάποιο σημαντικό αντίκτυπο σε ό,τι αφορά την κατανομή του εισοδήματος σε αυτή τη χώρα. Άρα λοιπόν μέσω της επιβολής κάποιων τέτοιων νέων νόμων κατέφερα, κατάφεραν οι ΗΠΑ την καλύτερη κατανομή του εισοδήματος. δηλαδή, ε, έφταναν οι φορολογικοί συντελεστέ σε ό,τι αφορά την κληρονομιά, όταν αυτή ήταν πολύ μεγάλη, στο 77%. Και εδώ δεν αναφέρομαι στη Σοβιετική Ένωση σε κάποιο άλλο καθεστώ, αναφέρομαι στι Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, δηλαδή ότι κατάφεραν με τέτοιου είδου νομοθεσία να, να, να φτάσουν σε μια λίγο πιο ισότιμη κοινωνία. Άρα λοιπόν, τέτοιου είδους νόμοι πράγματι μπορούν να αποτελέσουν τον καλύτερο τρόπο για να επιτύχουμε καλύτερη πιο ισότιμη κατανομή του εισοδημάτων στι κοινωνίε μας. Ένα τρίτο στοιχείο στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι η ανισότητα σε ό,τι αφορά αυτούς που έχουν μια θέση εργασίας και εκείνους που δεν έχουν μια θέση εργασίας. Αναφερθήκαμε εδώ στην τέταρτη επανάσταση, δηλαδή στην βιομηχανική επανάσταση καταρχήν με, την, με τον ατμό ε, και ούτω καθεξής. Ε, σε κάθε πάντως επανάσταση αυτό που ε, είδαμε ήταν μείωση του χρόνου εργασίας από 80 σε 60 και γύρω στα 1960 στο 48, στο 70 Στη δεκαετία του 70 φτάσαμε στις 40 και στις έχουμε φτάσει στις 38,5 με 35 ώρες εργασίας στις ε, πολύ ανεπτυγμένες ε, περιοχές. Οπότε γιατί δεν αναφερόμαστε και πάλι εδώ σε αυτή τη νέα επανάσταση στη μείωση των όρων εργασίων κάθε φορά όπου είχαμε ιστορικά αύξηση της παραγωγικότητας μέσω ακριβώς νέων εφευρέσεων, για παράδειγμα των ατμομηχανών, ε, τώρα εδώ με την ψηφιοποίηση, γιατί δεν μπορούμε και πάλι να κάνουμε λόγο στη μείωση των ορών εργασίας. Γιατί δεν κάνουμε λόγο για παράδειγμα για 30, 25 ε, ώρες εργασίας. Στην ε, Volkswagen ε, νομίζω ήδη εφαρμόζει τέτοιου είδου ώρες εργασία. Νομίζω σε, κάποιες, σε κάποια εργοστάσια είναι στι 30 ώρε, αν θυμάμαι καλά, χωρί να μειωθούν οι μισθοί. Αυτά λοιπόν ήθελα να πω από τον λόγο. Σας ευχαριστώ κυρίες και κύριοι θα μιλήσω για ένα κάπως διαφορετικό θέμα από ότι οι προλαλήσαντες. Πρέπει να καταλάβουμε κάτι, ότι σήμερα πρέπει να γνωρίζουμε όχι μόνο πώς οι αλλαγές στην κοινωνία την επηρεάζουν, αλλά πόσο αναλογικά λάβουμε κάτι. Ότι σήμερα πρέπει να γνωρίζουμε όχι μόνο πόσοι οι αλλαγές στην κοινωνία την επηρεάζουν, αλλά πόσο αναλογικούς αν θέλει να μειώσει κανείς τις κοινωνικές ανισότητες, απλώς τελικά οδηγείται σε διαφορετικό είδος ανισοτήτων. Ώρες όσον αφορά τον κοινωνικό αποκλεισμό, τη φτώχεια και άλλα προβλήματα. Όσον αφορά τη διαθεσιμότητα, η τσεχική δημοκρατία δεν έχει μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τις εσωτερικές ανισότητες. Σύμφωνα με τον ΟΣΑ, και στο 3%. Μηδέν είναι απόλυτη ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στους μισθούς. Στην Τσεχική Δημοκρατία λοιπόν είναι πολύ μικρές οι διαφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 0,27 είναι στη Σουηδία, στη Σλοβακία 0,25. Όσον αφορά τις ίσες ευκαιρίες και την κοινωνική ένταξη και συμπερίληψη, ένα από τα μεγαλύτερα θέματα στη Τσεχική Δημοκρατία είναι η ύπαρξη αποκλεισμένων περιοχών και περιφερειών. Και αυτό πηγαίνει μαζί με πολύ μικρή δυνατότητα να συμμετάσχουν οι κάτοικοι στην αγορά εργασίας, να έχουν καλή εκπαίδευση και να μπορούν να συμμετέχουν ε, στην κοινωνική και πολιτική ζωή. Γι' αυτό το λόγο έχουμε μια νέα στρατηγική από το 2014 με το 2020. Για τη φτώχεια έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα στην Τσεχία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Eurostat του 2016 σε σύγκριση με το 2008 ο κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού έχει μειωθεί. Ήταν 1,375 εκατομμύρια άνθρωποι, 1.375.000 άνθρωποι οι περισσότεροι οι γυναίκες επηρεάζονται περισσότερο τις, ε, από τους άντρες. Όσον αφορά τη φτώχεια, ο, ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι για τα νοικοκυριά με ε, άνεργους ε, κατοίκους. Κάτι παραπάνω, 50,25 κάτι τέτοιο. Και αυτό το ποσοστό έχει αυξηθεί στην Τσεχική Δημοκρατία και μεγάλος κίνδυνος υπάρχει για τις ε, ε, οικογένειες που δεν είναι πλήρης ή οικογένειες όπου δεν πληρώνει ε, εκείνος που θα έπρεπε τη διατροφή όταν έχει βγει το διαζύγιο. Αν θέλουμε να είμαστε φιλόδοξοι στην Τσεχία, στα πλαίσια στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020, πρέπει να φροντίσουμε ώστε να μειώσουμε κατά 100.000 τους ανθρώπους εκείνους που κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν τη φτώχεια μέχρι το 2020. Τις μονογονικές οικογένειες πρέπει να προσέξουμε και να δούμε τι γίνεται με τους γονείς. Υπάρχουν καλές συνθήκες. Διαφορά ε, στις αμοιβέ, ανισότητα αμοιβών. Μπορούμε να παρακολουθούμε κάποιους δείκτες. Οι περισσότεροι δείκτες εστιάζονται επί συγκρίσεως ποσοστών των πλουσιωτέρων ανθρώπων και των φτωχοτέρων ανθρώπων. Σύμφωνα με έρευνα που έγινε το 2015, από το 10% των φτωχοτέρων οικοκυριών. Ε, κυρίως ε, προσέχουμε τις ανισότητες αμοιβή, το συντελεστή που αφορά τις ανισότητες αμοιβή. Την τελευταία δεκαετία αυτός ο συντελεστής, ο συντελεστής παραμένει σταθερός. Εν συγκρίση με άλλες χώρες, η τσεχική δημοκρατία, όπως και πολλές βόρειες χώρες, σκανδιναβικές χώρες, έχει παρόμοια τιμή στους δείκτες. Είναι πολύ πιο χρήσιμο να εστιαστούμε όμως επί των διαφόρων ξεχωριστών κοινωνικών ομάδων όσων απασχολούμενους σήμερα. Για αυτούς τους ανθρώπους, τους αυτοαπασχολούμενους, υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές. Διαφορές όσον αφορά το εισόδημα. Όμως, στην τσεχική δημοκρατία η κατανομή του εισοδήματος είναι πολύ αναλογική. Και αυτό διότι υπάρχει πάνω σε αυτό. Δηλαδή, πόσο εισόδημα πρέπει να ανακατανεμηθεί, ούτω ώστε να έχουν όλοι τουλάχιστον παρόμοια εισοδήματα. Στην τσεχική δημοκρατία πρέπει κανονικά να ανακατανείμουμε περίπου το 1 πέμπτο. Νέων επίσης επιβραδύνεται και μακροπρόθεσμη ανεργία και αυτή με χαμηλότερους βαθμούς μειώνεται. Μέλλον θα πρέπει να λάβουμε πολιτικές ε, πρωτοβουλίες στα πλαίσια του κοινωνικού πυλώνα της Ευρώπης. Θα πρέπει